The President of Ireland. Ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Είναι μεγάλη μας τιμή να καλωσορίσουμε τον κύριο Χίγκινς, πρόεδρο της Ιρλανδίας. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Χίγκινς θα μας μιλήσει. Πριν του δώσω το λόγο, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα. που είναι παρόντες εδώ, ο Μέγας Δούξ Γκυγιόμ και η γυναίκα του Στεφανή του Λουξεμβούργου. Καλώς ήρθατε. Επίσης χαίρομαι που δίπλα του στο θεωρείο είναι η σύζυγος ε, του Προέδρου Χίγκινς. Κυρία Χίγκινς, καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, και τώρα το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας, κύριος Χίγκινς. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε Κουίν, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να απευθυνθώ στο σώμα σας, όπου συνεδριάζουν οι δημοκρατικά άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών των 27 κρατών μελών που σύντομα θα γίνουν 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επίτροπε Γκέγεν Κουίν, σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στο σώμα σας, όπου συνεδριάζουν από κοινού οι δημοκρατικά άμεσα εκλεγμένοι των πολιτών των 27 κρατών μελών, που σύντομα θα γίνουν 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας απευθύνομαι ως Πρόεδρος της Ιρλανδίας. Το νησί μας είχε πάντα στενή σύνδεση με όλα τα ευρωπαϊκά θέματα. Η χώρα μας είχε πάντα στραμμένο το βλέμμα προς τα έξω. Έχουμε πολύ ισχυρές συνθέσεις με τον πολιτισμό και τη γνώση της Ευρώπης σε όλες τις διάφορες μορφές από την αρχαιότητα. Είμαστε ένα έθνος που πάντα εκτιμούσε ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό ανά τους αιώνες, αλλά και τώρα που η Ιρλανδία για έβδομη φορά κατέχει την εναλλασσόμενη Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών κατά το 40ο έτος ε, ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μέσω των αρχαίων κελτικών ε, σχέσεών μας, μέσω της συνεχής επαφής μας με την ευρωπαϊκή γνώση ή μέσω της σύγχρονης ε, μόνιμης στήριξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς οι Ιρλανδοί ήμασταν Ευρωπαίοι στην συνείδησή μας και στην αποφασιστικότητά μας. Η Ευρώπη πάντα υπήρχε στο πνεύμα των Ιρλανδών. Στην γοηδελική μας γλώσσα η μυθολογία της Ευρώπης ήταν πάντα παρούσε και μερικά από τα σύγχρονα θεατρικά μας έργα θυμίζουν τη χρήση που κάναμε των κλασικών πηγών της ελληνικής και ε, ρωμαϊκής μυθολογίας στα γοηδελικά παράνομα σχολεία των φρακτών που προϋπήρχαν της ε, ε, διάδοσης της χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Η γοηδελική γλώσσα που προηγείται της αγγλικής είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από ευρωπαϊκούς μύθους, ιδιαίτερα από τους μεγάλους μύθους της θάλασσας και της περιπλάνησης όπως η Οδύσσια του Ομήρου. Στον τομέα της ε, λογοτεχνίας, οι λαοί της Ευρώπης είχαν πάντα σεβασμό για την ε, πολιτιστική πολυμορφία που συχνά βασίζεται σε μια κοινή μυθολογία. Όμως, στα θέματα της διανόησης και του πνεύματος προσπάθησαν να συμβάλλουν όσο μπορούσαν περισσότερο Ιρλανδοί. Έτσι, τον Ιούλιο του 1950, ο τότε Ιρλανδός Πρωθυπουργός John A. Costello μαζί με τον Ιρλανδό Υπουργό Εξωτερικών και αργότερα κάτοχο του ε, ε, Νόμπελ Ειρήνη και ιδρυτικού μέλου τη Διεθνού Αμνηστία Σον Μακμπράιντ, πήγαν στο Λουξέι Λεμπάν για να εορτάσουν επισήμω την ε, χιλιοστή τετρακοσιωστή επέτειο τη γέννηση ενό από του μεγαλύτερου Αγίου τη Ιρλανδία και τη Ευρώπη του Κολομπάνε ο Κολομπάνος μαζί με τον Άγιο ε, Γκόλ δημιουργήσαν κέντρα γνώσης, ε, εικονογράφησης, χειρογράφων, κοινότητες και μοναστήρια σε όλη την Ευρώπη από το βορρά της Ιρλανδίας μέχρι τον Μπόμπιο όπου και ε, απεβίωσε ο Κολόμπενες. Αυτό το πνεύμα ε, ηθαγένειας, όπως θα μπορούσε να ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως θα μπορούσε να βοηθήσει τους Ευρωπαίους που θέλουν να δώσουν σε αυτές τις δύο λέξεις, Ευρωπαϊκή και Ένωση, μια άλλη έννοια, μια έννοια ανάπτυξης ε, των ανθρώπων. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω σε αυτήν την Ευρώπη που έχει αφιερωθεί στους πολίτες, που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Αλλά κάτι ακόμη για την συνάντηση του Λουξοϊ Λεμπάν τον Ιούλιο του 1950. Όπως και κάποιες συναντήσεις της ε, πρόσφατης περίοδου, η πραγματική ημερήσια διάταξή της δεν ήταν αυτή που είχε δημοσιευθεί. Είχαν πει ε, ότι ήταν εκκλησιαστική αλλά εκόβει το μικρόφωνο του Πρόεδρου, δυστυχώ. Α, τώρα ξανά άνοιξε. Είχε διακηρυχθεί ότι ήταν ε, τον Ιούλιο του 1957 συνάντηση λοιπόν θρησκευτικού χαρακτήρα. Όπω είπα λοιπόν, όπω και μερικέ πρόσφατε συναντήσει για τι οποίε δεν θα αναφερθώ, η ουσιαστική ημερήσια διάταξη δεν ήταν η δημοσιευμένη είχε ε, διακηρυχθεί ότι θα ήταν θρησκευτικού χαρακτήρα. Ήταν εκεί και ο παπικός νούσιος στη Γαλλία, ο καρδινάλος Ρονκάλι που αργότερα ήταν, ε, έγινε ε, ο Πάπας Ιωάννης 23ος καθώς και ο επίσκοπος του Μπόμπιο αλλά ξέρουμε από τις εργασίες της διακεκριμένης ε, επιστήμονος ε, της Ορβόνης Μαγκερίτ ε, Μαρίντε Μποά που είναι μοντερνίστρια, γλωσσολόγος, φιλόσοφος και λεξογράφος ότι ο πραγματικός στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να διευκολύνει μια συνάντηση του Ρομπέρ Σουμάν που ήταν πρόσωπος εξωτερικών της Γαλλίας με άλλους που είχαν τις ίδιες απόψεις για αυτόν από μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες και που ήθελαν να ακούσουν και να δοκιμάσουν τη μεγάλη του ιδέα για την δημιουργία μιας ένωσης των χωρών της Ευρώπης. Ο Σούμαν που το γνώριζε, γνώριζε τις προσπάθειες της Ιρλανδίας, θύμισε τις ε, παλιότερες ε, ε, περιπλανήσεις των μοναχών και δήλωσε ότι ο Κολομπάνος θα έπρεπε να είναι ο προστάτης Άγιος όλων όσων επιδιώκουν να οικοδομήσουν μια Ενωμένη Ευρώπη. Αυτή η συνάντηση του Σουμάν και οι άλλες που ακολούθησαν με τη βοήθεια του Ζαμονέ που συμμετείχε ανταποκρινόταν, προσπαθούσε να αντιμετωπίσει πρόσφατα και τρομερά γεγονότα. Αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και το τονίζω σήμερα, ότι στην απάντησή τους αυτή αναγνώρισαν την τεράστια αξία και βασίστηκαν στην ε, πλούσια γνώση της φιλοσοφίας, της ηθικής και της γενικές τάσης της ευρωπαϊκής σκέψης και δεν προσπάθησαν απλώς να αντικαταστήσουν τον πόλεμο Μερίνη, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, να δημιουργήσουν ένα όραμα, όραμα για τους λαούς της Ευρώπης που να συνεργάζονται χωρίς αποκλεισμούς. Δεν ήταν μια αφηρημένη προσπάθεια. Ήταν συγκεκριμένες προτάσεις, διανοητικές αλλά και με καρδιά για να ενωθεί η οικονομία και η ηθική ως προοπτικές για μια κοινή Ευρώπη για όλους αλλά η έμπνευση και τα επιτεύγματα των ιδρυτών πατέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι που πάντα θα ισχύει. Σήμερα οι πολίτες στην Ευρώπη απειλούνται από μια συνείδητη ροπή προς διχόνοια. Υπάρχει έλλειψη κοινωνικής συνοχής, ε, επανεμφάνιση του ρατσισμού και ένα αυξανόμενο έλλειμμα δημοκρατικής λογοδοσίας σε ε, μερικές αποφάσεις οικονομικού και χρηματοπιστωτικού είδους. Αυτά τα πληθυντικά σύννεφα κρέμονται πάνω από μια Ευρώπη που σε πιο ευτυχείς καιρούς είχε διαλέξει να βασίσει τον ύμνο της όχι σε κάτι σύγχρονο αλλά στο ποίημα του Φρίντριχ Σίλα «Ύμνο στη χαρά» και στη μελοποίησή του από τον Λούντβιχ Φαν Μπέιτοβεν στην ένατη συμφωνία. Τα κοινοβούλια έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν και πρέπει να συνεχίσουν να τον παίζουν αυτόν τον ρόλο. Αιώνες προσπαθειών έχουν γίνει από τους πολίτες της Ευρώπης για να κατακτήσουν την ψήφο για παράδειγμα για να επεκτείνουν σε όλους την ψήφο οι πολίτες προσβλέπουν στα κοινοβούλια για λογοδοσία έλεγχο, στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις εάν τα εθνικά κοινοβούλια το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να εγγυώνται τον έλεγχο πού θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η δυνατότητα υπάρχει εναλλακτική λύση που να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της συμμετοχικής δημοκρατίας δεν το νομίζω. Τα κοινοβούλια πρέπει να βασιστούν στην πείρα, στην ε, κληρονομιά της γνώσης, σε όλες τις, τις μορφές και πάνω απ' όλα στην καλύτερη, σύγχρονη, διανοητική εργασία και επιστημονική εργασία με πλουραλιστικό τρόπο. Έχω πλήρη συνείδηση σε αυτό το έτος ε, του Ευρωπαίου Πολίτη ότι ως κοινοβουλευτικοί είστε το εκλεγμένο συστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλεγμένοι από τους πολίτες από τόσο διαφορετικά εκλογικά σώματα που ψήφισαν στις ίδιες περίπου μέρες. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και στη συνεργασία σας με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ιδιαίτερα στο διάλογό σας με το εκλογικό σώμα, τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτοί οι πολίτες εμπιστεύονται εσάς όταν ψηφίζουν και σωστά έχουν προσδοκίες τα κοινοβούλια να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Καλωσορίζω ιδιαίτερα την αύξηση επιρροής και δυνατότητας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει κερδίσει, για παράδειγμα, για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές. Ήταν μια εξουσία που δεν την είχε το Κοινοβούλιο όταν σας επισκέφτηκα ως πρόεδρος και ε, προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού του 1996. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκτέλεση αυτής της ευθύνης εκ μέρους των πολιτών της Ευρώπης. Πώς θα είχαν αντιδράσει οι ιδρυτές της Ευρώπης στις ε, σημερινές ε, προκλήσεις. Ξέρουμε πόσο σκληρά εργάζονται οι θεσμοί για να ξεπεράσουν την πιο σοβαρή οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ένωση από την ίδρυσή της. Πόσο αγωνίστηκαν να αντιδράσουν αρκετά σύντομα να αντιδράσουν αποτελεσματικά στην τόσο σκληρή πρόκληση. Στην τόσο σκληρή πρόκληση που του απευθύνουν ε, πηγέ που δεν λογοδοτούν σε κανέναν. Δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονό ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε υποφέρουν από τα αποτελέσματα ενεργειών οργανισμών όπω οι οργανισμοί αξιολόγηση που αντίθετα από τα κοινοβούλια δεν λογοδοτούν σε κανέναν. Πολλοί από του πολίτε μα στην Ευρώπη θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της κρίσης ε, είναι αποσπασματική, κάποτε καθυστερημένη, δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα των καθηκόντων και συχνά ότι δεν επιδεικνύουν αυτές οι απαντήσεις σε επαρκή αλληλεγγύη με αυτούς στις απειλές που υφίστανται ή στις ε, πραγματικές οικονομικές δυσχέρειες που υφίστανται. Θεωρούν ότι γενικά η οικονομική κυρίαρχη σκέψη των πρόσφατων ετών βασίζεται σε στεγνές τεχνικές αντιλήψεις. Για παράδειγμα, υπολογισμούς που είναι αφηρημένοι, δεν βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα όπως η ανεργία, που κυρίως ενδιαφέρονται γιατί οι επιπτώσεις θα έχουν τα μέτρα στις κερδοσκοπικές αγορές, αντί να ενδιαφέρονται και να βασίζονται σε επαρκή συμπόνια και κατανόηση για τα προβλήματα των πολιτών της Ευρώπης που είναι όλοι μέλη μιας ένωσης και για τους οποίους πολίτες όλοι, όλοι οι πόροι της Ευρώπης, πολιτική, κοινωνική, οικονομική και διανοητική, θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί εάν η Ένωσή μας είχε ως βάση μια ηθική προοπτική. Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανεργία, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε μόνο και αποκλειστικά ένα μόνο ηγεμονικό πρότυπο που να εξαιρεί όλα τα άλλα, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματά μας όπως η ενεργεία. Δεν μπορούμε ε, τυφλά να αποδεχόμεθα μια πρακτική οικονομική θεωρία με πολύ στενή βάση και υποθέσεις, με μια βάση που ε, είναι αμφισβητήσιμη και που δεν ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων που προτείνει. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρούνται απλώς μια οικονομική περιοχή όπου αντιμάχονται οι ισχυροί τους αδύνατους. Οι πολίτες μας ε, επιθυμούν μια γνώση, μια γλώσσα αλληλεγγύης. Θέλουν να υπάρχει συνοχή, θέλουν να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε ένα μέλλον ειρήνης, ευημερίας, όπου να συμμετέχουν όλοι μια Ευρώπη της δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση. Γιατί αν αποτύχουμε υπάρχει κίνδυνος η οικονομική κρίση να οδηγήσει σε κρίση νομιμοποίησης της Ένωσης. Στις ε, ιδρυτικές της συνθήκες η Ένωση βασίζεται σε αξίες όπως ο σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζει την νόμιμοποίησή της στην στήριξη των πολιτών. Αυτή η σύνδεση με τους πολίτες, αυτή η πίστη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από αυτούς και για αυτούς, είναι θεμελιώδης. Χωρίς αυτήν δεν έχουμε ε, έρισμα και οι πολίτες χρειάζονται να απευθυνόμεθα και στην καρδιά και στο πνεύμα τους. Χρειάζονται διαβεβαιώσεις ότι η Ένωση θα τηρήσει τις ε, ιδρυτικές συνθήκες. Πριν από μερικά χρόνια η Ευρώπη είπε ότι η Ευρώπη, ε, ο Ζακ Ντελόρ είπε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ψυχή. Αλλά αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε κληρονόμοι μιας πολύ σημαντικής ε, βάσης ευρωπαϊκών αξιών. Η ελληνική δημοκρατία, το ρωμαϊκό νομικό σύστημα, η, ευρω, η, η χριστιανική παράδοση, ο προτεσταντισμός, ο διαφωτισμός, η μεγάλη δημοκρατική επανάσταση που ξεκίνησε στη Γαλλία. Η Ευρώπη δεν είναι απλώς λοιπόν χώρος ε, οικονομικών ανταγωνισμών όπου οι πολίτες μας θα πρέπει να θυσιάζουν τη ζωή τους σε ένα ε, αφηρημένο πρότυπο οικονομίας και κοινωνίας που δεν έχει βασιστεί σε εκλογική νομιμοποίηση. Κοιτάζοντα προ το μέλλον, πρέπει να βασιστούμε σε αυτέ τι ιδρυτικέ αξίε τη Ένωση, που συμπεριλαμβάνουν την συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ των πολιτών τη Ένωση και μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του υπόλοιπου κόσμου. Πρέπει να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε από κοινού ένα καλύτερο μέλλον. Όπω είπε και ο Ζακ Ντελόρ, για την σημερινή κρίση. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο πυροσβέστες, χρειάζεται και αρχιτέκτονες. Ένα πρώτο και πήγον καθήκον είναι η Ευρώπη να επανέλθει σε βιώσιμη και ουσιώδη απασχόληση και να επανέλθει σε ουσιώδη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο διαβροτικό για την κοινωνία και πιο συντριπτικό για τους πολίτες παρά η ε, εμένουσα ανεργία, ιδιαίτερα για τους νέους. Αυτή τη στιγμή 26 εκατομμύρια πολιτών σε όλη την Ένωση είναι χωρίς εργασία. 5,7 εκατομμύρια εξ αυτών είναι νέοι και 115 εκατομμύρια στην Ένωσή μας κινδυνεύουν από την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οι Ιρλανδικές Προεδρίες πάντα βασίζονταν στο πνεύμα των ιδρυτικών συνθήκων. Η παρούσα Ιρλανδική Προεδρία γι' αυτό έχει θέσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας ως πρώτη προτεραιότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η αντιμετώπιση τη ανεργία είναι η πιο σημαντική κοινωνική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Στην ε, κοινωνική συνάντηση κορυφή του περασμένου μήνα, σωστά προειδοποιήσατε για τι επιπτώσει ε, τη εξάπλωση τη ανεργία και τη φτώχεια στην Ευρώπη. Γι' αυτό επενώ την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Φεβρουάριο για την πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων και τι προτάσει τη Κομισιόν να αρχίσει να λειτουργεί στην αρχή του επόμενου έτους. Είναι επίγον το θέμα αυτό και καλωσορίζω και τη συμφωνία που επιτέχθηκε στο Συμβούλιο για το πρόγραμμα εγγύσεων για τους νέους που θα διασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι 125 θα έχουν μια καλή προσφορά εργασίας, εκπαίδευσης, μαθητείας ή κατάρτισης ε, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που γίνονται άνεργοι. Αλλά πρέπει να κάνουν περισσότερα. Πρέπει και οι γυναίκες να συμμετέχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας. Οι γυρεότεροι εργαζόμενοι να μην μένουν στο περιθώριο και ότι οι μακροπρόθεσμα άνεργοι να έχουν ε, πλήρω τα προσόντα που χρειάζονται για να επανέλθουν στην εργασία. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχασαν τη δουλειά τους δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή ιδιαίτερα στην πολιτιστική πλευρά των κοινοτήτων τους. Πρέπει επίση να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να, να ευνοήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά πολλών κοινοτήτων. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους αυτούς και για άλλους. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την δημιουργικότητα, την καινοτομία, το επιχειρηματικό πνεύμα. Μια γενναιόδωρη λοιπόν προοπτική για την Ευρώπη, ένα γενναιόδωρο όραμα. Δεν κοιτάζει μόνο προ το εσωτερικό. Το ευρωπαϊκό πρότυπο έχει εμπνεύσει πάρα πολλού στην προσπάθειά του για ειρήνη και δημοκρατικού θεσμού. Και ναι, μεν μπορεί ο πυρσό τη αυτή τη στιγμή να μην λάμπει τόσο λαμπρά, αλλά παρόλα αυτά η Ευρώπη μπορεί να γίνει φάρο ελπίδα και ενθάρρυνση για πολλού λιγότερο Ευτυχεί ανθρώπου στον κόσμο. Εάν είμαστε ενωμένοι για το, την κλιματική αλλαγή, αν αναγνωρίζουμε ότι αυτοί που λιγότερο συμμετέχουν στα σφαιρικά μα, στα πλανητικά μα προβλήματα πληρώνουν την υψηλότερη τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα κάνουμε κάτι σημαντικό. Εμεί είμαστε ο μεγαλύτερο δωρητή τη προσπάθεια κατά τη πείνα και, και ε, του υποσυντισμού. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βοηθάει τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένα σημαντικό τεστ για το κύρος τη και την αξιοπιστία τη. Θα επιτρέψει η Ένωση οι τωρινέ οικονομικέ τη διχείρε να υπονομεύσουν τη δέσμευσή τη για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα πλανητικά προβλήματα, ο, η πείνα, η φτώχεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κλιματική αλλαγή. Ελπίζω όχι. Θα πρέπει να επαναβεβαιώσουμε το γενναιόδρο ιδεαλισμό που είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού οράματο για αντιμετωπίζοντα εκ νέου αυτά τα προβλήματα αλληλέγγυα με του εταίρου μα. Ελπίζω ότι θα το κάνουμε διότι τα μέτρα που θα ε, είναι η συνέχεια των, στόχων, των αναπτυξιακών στόχων της ε, χιλιετίας, πώς θα σεβαστούμε την πολυμορφία, τους διαφόρους, διαφορετικούς δρόμους προς την ανάπτυξη με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο τους, θα είναι ένα μεγάλο τεστ για την ευρωπαϊκή κοινότητα και τον πλανήτη. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει το καθήκον να αντιμετωπίσει και το παρελθόν τη, ιδιαίτερα τι πιο ζωφερέ περιόδου τη αυτοκρατορία, με ειλικρίνεια και το μέλλον τη με δέσμευση για τι αρχέ που είναι κοινέ σε όλη την ανθρωπότητα, με ένα λόγο που σέβεται την πολυμορφία, μπορεί να συμβάλλει ουσιοδέστατα. Όχι μόνο για του πολίτε τη ίδια τη Ευρώπη, αλλά για όλου του ανθρώπου. Μπορεί να είναι ηγετική στη δημιουργία μια ε, ηθικής που αναγνωρίζει τις ευθύνες από γενιά σε γενιά. Μια τέτοια ενοποιημένη προσπάθεια, πρέπει να το πω ειλικρινά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η βασική η υπερέχουσα προσέγγιση μοιάζει να βασίζεται σε έναν τρόπο σκέψης που δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσει, που δεν είναι σε θέση ή και που είναι απρόθυμη να ξεφύγει από αυτό το στενό τρόπο σκέψης. Και αν εμείς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις. Υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε μια ηθική και διανοητική αδυναμία δράσης. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στην ε, ε, ριζοσπαστική σκέψη και στην κληρονομιά σε αυτό το τομέα από το παρελθόν. Στην κοινή διανοητική μας κληρονομιά έχουμε πολλά στα οποία θα μπορούσαμε να βασιστούμε. Ας θυμηθούμε ότι στα πλαίσια της ε, νέας σκέψης που για παράδειγμα ήταν το χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού διαφωτισμού που είχε βασιστεί αυτός ο ίδιος σε παλιότερους αρχαίους διαφωτισμούς υπήρχαν σημαντικά παραδείγματα διαφωνούντων και ριζοσπαστικών. Α μην ξεχνάμε ποτέ τα ιδιαίτερα παραδείγματα που μας δίνουν αυτοί οι διαφωνούντες στοχαστέ Ντενί Διδγό, Ιμάνιουλ Καντ και ο Χέρντερ. Αυτοί στην εποχή τους βρήκαν τα μειονεκτήματα του διαφωτισμού που ήταν υπέρ της αυτοκρατορίας και του υπεριαλισμού και με τα βιβλία τους, τα φυλάδια τους και τους λόγους τους αμφισβήτησαν αυτή τη λογική αυτή η καθαρά πρακτική οικονομική σκέψη που αυτή τη στιγμή είναι το ηγεμονικό μοντέλο της οικονομικής θεωρίας όχι μόνο στην Ευρώπη είναι το μειονέκτημα των καιρών μας. Αυτή η νεοκλασική οικονομική σκέψη που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι φυσικά χρήσιμη για κάποια περιορισμένα και σωστά καθορισμένα προβλήματα. Είναι ανεπαρκής ωστόσο ως προσέγγιση για τα μεγαλύτερα προβλήματά μας και το μέλλον μας. Χρειαζόμαστε νέα, ουσιώδη, πλουραλιστική, πολιτική και οικονομική σκέψη και έναν λόγο απελευθερωτικό που να τους εκφράσει. Και θεωρώ ότι αυτά είναι δυνατά, διότι το κυρίαρχο μοντέλο και η μέθοδό του, η μέθοδός του δεν καθορίζει μόνο το λόγο, αλλά και τις πολιτικές επιλογές. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη για νέα μοντέλα σύνδεσης μεταξύ της οικονομίας, της κοινωνίας και των πολιτικών που αποφασίζουμε. Αυτό είναι ουσιαστικό για ουσιοδό πλουραλιστικέ επιλογέ στι πολιτικέ μα, αλλά βεβαίω και για δημοκρατική λογοδοσία και ουσιώδου σχέση με τα ουσιαστικά μα προβλήματα. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τι ε, παρούσε προκλήσει, εσεί ω Ευρωπαίοι κοινοβουλευτικοί σα καλώ να επιτρέψετε τα νέα αυτά μοντέλα στον ευρωπαϊκό λόγο. Να του δώσετε τη δυνατότητα να εκφραστούν στο κοινοβούλιο σα και στα άλλα θεσμικά οργάνα τη Ένωση. Για να επιτύχουμε αυτό το λόγο, ο ρόλος των διανοωμένων είναι πολύ σημαντικός. Των διανοωμένων που συμμετέχουν στην, ε, στον πολιτικό διάλογο. Θα πρέπει να πούν δημοσίω και κατηγορηματικά ότι τα προβλήματα της Ευρώπης δεν είναι απλώς τεχνικά και δεν μπορούν να επιληθούν μόνο με τεχνοκρατικές λύσεις χωρίς να υπάρχει δημοκρατική λογοδοσία. Ορισμένοι ισχυρισμοί ότι οι πολίτες και οι εκπρόσωποι τους δεν έχουν επαρκείς ε, χρηματοπιστωτικές και οικονομικές γνώσεις για να εφαρμόσουν τις αναγκαίες αποφάσεις για πολιτικές που αφορούν τις ζωέ τους, για την ανεργία δηλαδή, για την στέγαση, την ε, υγεία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον, έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά την νομιμοποίηση των ενεργειών μας. Πρόκειται για ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ίδια τη δημοκρατία. Ένα άειλο, μία άειλη μορφή του οικονομικού χώρου υποκαθιστά τους λαούς, τις κοινωνίες και τα κράτη. Χάνει την επαφή με την ιστορία και τους, τις σύγχρονες προκλήσεις και δεν έχει την ηθική σύνδεση με την ηθική και την αλληλεγγύη που χρειαζόμαστε. Μια τέτοια οικονομική σκέψη αποφεύγει και δεν αντιμετωπίζει τις παρούσες προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πρόκειται να γίνει σεβαστή όπως το μεγάλο όραμα που είναι και πρέπει να είναι, πρέπει να βασιστεί στην πολιτιστική κληρονομιά και τα ταλέντα και τις δυνατότητε των λαών της Ευρώπης. Αυτή θα είναι μια πραγματική ένωση, εάν κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ελεγγύη. Καταλήγοντας, εάν η Ευρωπαϊκή μας Ένωση και οι προοπτικές δεν είναι αυτού του ουσιώδους χαρακτήρα, πρέπει να γίνει τώρα με αλλαγές στην συνειδητοποίηση και τη δέσμευσή μας, με επαναβεβαίωση του ιδεαλισμού, του ηθικού μας θάρρους, και τη διανοητική ισχύω που ήταν η βάση των ε, ενεργειών των ιδρυτικών πατέρων της Ευρώπης. Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη είναι λαοί με ιστορία, με ανάγκες και με κοινέ δυνατότητε. Εάν εναλλακτικά θεωρούμε ότι οι λαοί μα είναι απλώς μεταβλητέ ε, ε, στις εξισώσεις των οργανισμών αξιολόγηση που δεν λογοδοτούν σε κανένα δήμο και που επανειλημμένα έχουν σφάλει, τότε αντί να είμαστε πολίτε, θα γίνουμε απλοί καταναλωτές. Πιόνια στην κερδοσκοπική σκακέρα χρηματοπιστωτικών κινήσεων σε ένα παιχνίδι που βασίζεται σε υποθέσεις που είναι αδύναμες, που δεν έχουν ελεγχθεί και πολύ συχνά ούτε καν ομολογημένες. Θέλω λοιπόν οι αποφάσεις μας να έχουν επιπτώσεις, να μην είναι απλώς στενά τεχνοκρατικές. Αυτό δεν είναι απλώς χρήση των διανοητικών μας δυνατοτήτων. Είναι για να υπερασπιστούμε και να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία. Αναγνωρίζω βεβαίω και θέλω να είμαι πολύ σαφή. Πιστεύω πάρα πολύ στη χρησιμότητα σε πολλούς τομείς των πρακτικών οικονομικών. Όμως πιστεύω ότι εάν οι μέθοδοι αυτών των οικονομικών υποκαταστήσουν την ολοκληρωμένη, ενοποιημένη, πολυθεματική γνώση που τώρα χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά πλαίσια και τις ανάγκες των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, εάν λοιπόν βασιστούμε αποκλειστικά σε μια τόσο τεχνοκρατική προσέγγιση, θα είναι ανεπαρκή η απάντησή μα. Εάν θέλουμε με Ευρωπαϊκή Ένωση ειρήνη και ενημερία, όπω την ήθελαν οι ιδρυτέ μα και που πιστεύω την θέλουν οι πολίτες της Ευρώπης πέρα από τον κατανοητό φόβο των ε, τρεχουσών περιστάσεων, εάν θέλουν μια στρατηγική που να βασίζεται στην έρευνα, τη γνώση και τι απόψει όλων των κοινωνικών επιστημών, τη ηθικής και τη φιλοσοφία. Αυτό χρειαζόμαστε. Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτέ, υπουργοί, επίτροποι, από τις διαφορετικές μας ιστορίες, από τα προβλήματά μας, από τους φόβους και τις προσδοκίες μας. Ελπίζω ότι θα προκύψει μία αντίδραση που θα αποτελέσει ένα πολύχρωμο, ένα ε, χαλί που θα έχει διαφορετικά ε, χρώματα που θα βασίζεται στην ε, μνήμη και στις ε, επιτυχίες του πνεύματός μας. Δεν έχει σημασία τελικά εάν θα είναι οι ελπίδες μας ή καθαρά η γνώση μας. Αλλά όλα αυτά πρέπει να συμμετάσχουν όλα μαζί με, να συνεργαστούμε με ε, ανοιχτό τρόπο προς τον κόσμο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και τις μέλους της γενιάς, να βοηθήσουμε όλο το λαό μας ισότιμα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν εμείς οι πολίτες της Ένωσης που θέλουμε να υπάρξει μια πραγματική ένωση, να βγούμε από το σκότος προς το φως, να επιτύχουμε κάτι που να είναι όντως αντάξιο του ποίηματος του Σίλερ που αρχικά είχε ως τίτλο «Οδή προς την ελευθερία». Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Χιγγένς. Εξαιρετική η ομιλία σας. Δεν ξέρω αν είναι όλοι εδώ, έχουν την ίδια άποψη μαζί με τη δική σας. Εγώ πραγματικά σας άκουσα με μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν ξέρω αν όλοι το σκέφτηκαν το ίδιο αλλά ένα μπορώ σίγουρα να σας ε, πω. Ε, η Ιρλανδία πραγματικά είναι ευτυχής χώρα με έναν εξαιρετικό πρόεδρο σαν, σαν εσάς. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η ομιλία σας και μας δώσατε πάρα πολύ θάρρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.